Είναι Ολομέλεια λαμβάνει χώρα στις 25 Νοεμβρίου από τις 9 ως τις 1 και από τις 3 ως τις 7. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό ύπνο σε όλους.